αφορά τον κύριο Ρίμουν Σερνατζότο, ο οποίο φεύγει από την ομάδα του ΕΛΚ και θα μεταβεί στην ε, ομάδα του ECR από σήμερα, 7 Ιουλίου. Επόμενη